Κυρίε uh, I'm very... Κυρίε και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Ξεκινήσω εγώ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα λίγο να ξεκινήσω, αλλά είχε να κάνει με τη διαδικασία στην Ολομέλεια. Επιτρέψατε μου να σας καλωσορίσω σε αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω σύθιστε ότι η συνεδρίασή μας ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο και έχουμε διερμηνία στις ε, στις γλώσσες των πλήρων μελών της ε, υποεπιτροπής. Αυτό είναι μια προτεραιότητα. Επιτρέψατε μου λοιπόν να προχωρήσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης που είναι πολύ απλή. Τη απουσία παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου επίσης να ζητήσω συγγνώμη για τις ε, αλλαγές στην Προεδρία, στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, διότι που οφείλονται σε σημαντικές συζητήσεις στην ε, αίθουσα της ε, Συνόδου της Ολομέλειας και θα πρέπει να εναλλασσόμεθα η Προεδροί. Μετά από λίγο λοιπόν θα με αντικαταστήσει ο κύριος Στέτινα και ίσως και ακόμη κάποιος άλλος αντιπρόεδρος. Γιατί και ο κ. να συμμετέχει στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας μας διάταξης. Ε, επιτρέψατε μου να καλωσορίσω εξ ονόματος όλων των εξέχοντα προσκεκλημένων μας είναι η συνέχεια της δικής μου και της δικής σας επίσκεψης στην, στο στρατηγείο του Eurocorps και έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε σήμερα τον αντιστράτηγο Αλφρέντο Ραμίρες και τον ταξίαρχο Franz Χαβέρ Είναι η εμπειρία τους στην Eurocorp που παρέχει την σταθερότητα και την ειρήνη σε πολλές περιοχές του κόσμου και υπάρχει επίσης κάποια πρόοδος στην συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ μάθαμε ότι η δήλωση και το μνημόνιο που είναι ο επικεφαλής και διευθυντής του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προοδεύσει Επιπλέον, ο ταξίαρχος Φρέγκλε έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τη δική μας συζήτηση, διότι το επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αποστολής Κατάρτισης στο Μαλί του EUTM Ε, για το οποίο θα συζητήσουμε στο επόμενο εξάμεινο φέτος. Χωρίς περισσότερη λοιπόν καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο και να καλωσορίσω θερμά τον αντιστράτηγο Αλφρέντο Ραμίρες και μετά τον ταξιερχό Φράντσι Χαβιέρ ε, Φρέγκλε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Okay. Ε, ε, Καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας πόσο μας τιμά η πρόσκλησή σας σε αυτήν την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι αντιστράτηγος, ο αντιστράτηγος Αλφρέντο Ραμίες, επικεφαλής του Eurocor. Και εδώ αριστερά μου είναι ο ταξίαρχος Φραντς Φρέγκλεϊ, που είναι επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του Eurocore. Θα επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα κύρια θέματα που κατά τη γνώμη μου εξηγούν τι είναι και τι κάνει το Eurocore. Ιδιαίτερα θέλουμε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πέντε χώρες που συμμετέχουν στο πλαίσιο του Eurocore προσπαθούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ του Eurocore και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πιο πρόσφατες και μελλοντικές μας δραστηριότητες για την υπεράσπιση της Ευρώπης. Στα πλαίσια των αμυντικών μας δραστηριοτήτων και μετά ο ταξίαρχος Φρέγκλε, ο επικεφαλής του Γενικού μας Επιτελείου, θα σας ε, εξηγήσει πώς πήγε η αποστολή μας UTM. Τονίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίζεται η συνολική ασφάλεια. Αυτό είναι όλο και πιο περίπλοκο και πρέπει να έχουμε τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Τα ευρωπαϊκά προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις. Το βασικό πλαίσιο που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη ε, αστάθεια και αβεβαιότητα. Γύρω μας υπάρχει ένα τόξο αστάθειας από το Σαχέλ στο Νότο μέχρι τα ανατολικό μας σύνερα, περνώντας από τη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο. Η διασύνδεση και διαφορετικότητα αυτών των απειλών σημαίνει ότι δεν είναι μόνο στρατιωτικού χαρακτήρα, αλλά και κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού. Όλα αυτά μαζί όπως αποδεικνύουν και τα τελευταία γεγονότα, η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης σημαίνει ένα σύνολο μέσων που ε, υπερβαίνει την απλή στρατιωτική ανταπόκριση. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ εδώ και μερικούς μήνες, η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα ήπια δύναμη. Αλλά συνέχισε λέγοντας, αλλά ακόμη και οι πιο ισχυρές ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να δράσουν μακροπρόθεσμα εάν δεν έχουν τουλάχιστον κάποιες ε, ολοκληρωμένες, ενοποιημένες δυνατότητες άμυνας. Για να συμβάλλουμε στρατιωτικά σε αυτήν την περίπλοκη κατάσταση οι μονάδες μας αποτελούν την πιο κατάλληλη οργανωτική δομή που μας παρέχει όλες τις δυνατότητες για να δράσουμε αποτελεσματικά από τη δημιουργία του. Το Eurocore είναι η απόδειξη ότι είναι δυνατόν να υπάρξει αποτελεσματική πολυεθνική συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Έχει χαρακτήρα τμήματικό που του επιτρέπει να λειτουργεί ε, με διάφορες μορφές. Θέλουμε λοιπόν το γενικό μας επιτελείο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα κρίσεων που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Ένωση. Είμαστε πεπισμένοι ότι το Eurocore εξακολουθεί να είναι και σήμερα η καλύτερη ανταπόκριση την κατάλληλη στιγμή στις διαδικασίες που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή κατάσταση. Το Eurocore μπορεί να είναι λοιπόν πρότυπο μια σταδιακής ενοποίησης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων, ε, ενόπλων δυνάμεων. Και χαιρόμεθα που μπορούμε να είμαστε πρότυπο και ορισμένοι ακριβώς ε, μας χαρακτηρίζουν πρότυπο από την ίδρυσή του. Το Eurocore είχε πάντα και μια πολιτική διάσταση. Το γενικό μας επιτελείο σταδιακά έχει αποκτήσει και ευρεία νομιμοποίηση και πείρα και έχει διτό χαρακτήρα. Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ κάτι που το καθιστά μοναδικό. Όταν η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει νέες, νέες αλλά και παλιές απειλές και κινδύνους το Eurocore είναι στη διάθεσή της για να αξιοποιηθεί ως στρατιωτικό όργανο για να ενισχύσει την ασφάλεια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας αξιοποιώντας έτσι την εμπειρία μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Eurocore πρέπει να το γνωρίζουν οι ηγέτες ε, της Ευρώπης, η πολιτική και η στρατιωτική. αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ και σας παρουσιάζω το Eurocore και κατά τη διετή θητεία μου έχω καθορίσει μεταξύ των καθηκόντων μου και μάλιστα ε, ως μία από τις προτεραιότητες μου να γίνει γνωστό το Eurocore για να είναι ακριβώς η στρατιωτική δύναμη που θα πρέπει να προτιμάται για οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το 1992 από τη Γαλλία και την Γερμανία. Αλλά είχε από την αρχή σαφή ευρωπαϊστική κατεύθυνση. Εξακολουθεί να είναι ένα εργαλείο και πολιτικό και στρατιωτικό. Όλοι καταλαβαίνουμε την συμβολική αξία του ότι το γενικό μας επιτελείο και το στρατηγείο μας είναι εδώ στο Στρασβούργο που είναι σύμβολο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, στην καρδιά της Ευρώπης. Από τότε που 2009 που άρχισε να ισχύει η λεγόμενη συνθήκη του Στρασβούργου, το Eurocore έχει σαφή και οριστικό πολυεθνικό χαρακτήρα. Η λήψη αποφάσεων βεβαίω σε ένα πολυεθνικό πλαίσιο είναι πιο περίπλοκη, αλλά αποδίδει και μια νομιμοποίηση που την καθιστά απαραίτητη. Νομιμοποίηση και πολυεθνικότητα. Πάνε χέρι με χέρι. Εδώ στην οθόνη βλέπετε τις πέντε χώρες ε, από τις οποίες απαρτίζεται το Eurocore. Και αν όλα πάνε καλά η Πολωνία θα είναι η έκτη χώρα που θα ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό τον επόμενο Ιανουάριο. Εξαρτώμεθα βέβαια από τα γενικά επιτελεία των πέντε χωρών που ε, απαρτίζουν το Eurocore. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πιο ψηλό επίπεδο και πάντα ομόφωνα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ σε αυτή τη διαφάνεια ότι οι πέντε συν μία χώρες αποτελούν πάνω από 50% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες τρεις χώρες συμβάλλουν στο στρατηγείο μας ως ε, συνδεδεμένα μέλη, έτσι τις αποκαλούμε. Αυτό ε, διευρύνει ακόμη περισσότερο την πολυεθνικότητά μας. Σε μερικές εβδομάδες, τέλη Μαρτίου, προβλέπεται ότι και η Ρουμανία θα είναι το τέταρτο συνδεδεμένο μέλος. Έχει ήδη επικυρωθεί. Όπως θα δείτε λίγο παρακάτω, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ενταχθούν και άλλα κράτη σε αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε μια διάσκεψη, θα αναφερθώ παρακάτω, τον προσεχή Απρίλιο, για να αυξήσουμε τα κράτη-μέλη μας. Και είμαι πλήρως πεπισμένος ότι το κύριο χαρακτηριστικό του Eurocore είναι ο γνήσια πολυεθνικός του χαρακτήρας. Αυτό του δίνει κρίσιμα πλεονεκτήματα. Όταν το 1992 δημιουργήθηκε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά στην πραγματικότητα το στρατηγείο μας έχει συμμετάσχει τέσσερις φορές σε πάντα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό μας δίνει πολύ, πολυεθνική πείρα που είναι η βάση της αξιοπιστία μας, ιδιαίτερα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, όπως βλέπετε εδώ, για πρώτη φορά αναπτυχθήκαμε στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη το 1998, το 2000 στο Κοσφοπέδιο, 4 και 5 στο Αφγανιστάν, στα πλαίσια του ΙΣΑΦ και το 12 επίσης στα πλαίσια του ΙΣΑΦ και δύο φορές ως NAF, ε, δύναμη ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ. Έχουμε αυτόνομο χαρακτήρα και είμαστε διτεθειμένοι να αναπτυχθούμε ταχύτατα. Λοιπόν, αυτά για το παρελθόν. Να σας μιλήσω τώρα για το παρόν. Εδώ βλέπετε τις ε, λειτουργικές μας δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια. Όπως βλέπετε, εστιάζουμε σε αυτά στο οποία εστιάζει και έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περασμένο καλοκαίρι αναπτυχθήκαμε στα πλαίσια του EUTM στο Μαλί. για να εκπαιδεύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του στα πλαίσια του ταξιάρχου Φρέγκλε που ήταν επικεφαλής της αποστολής και θα σας μιλήσει μετά για να σας δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτή την αποστολή. Επίσης το δεύτερο εξάμεινο του 16 το Eurocore θα αναλάβει το ρόλο του στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ομάδας Μάχης, της Ομάδας Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Battle Group. Θα κάνουμε διάφορες ασκήσεις για να λάβουμε την τελική πιστοποίηση ότι είμαστε ομάδα μάχης ε, τέλη του χρόνου. Και το επόμενο βήμα θα είναι να είμαστε εμείς το πρώτο εξάμεινο του 17 ακριβώς το στρατηγείο. Δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 16 και το πρώτο του 17 θα έχουμε αυτές τις δραστηριότητες. Και εντωμεταξύ το Eurocore έχει δυνατότητα να συμμετάσχει και σε άλλες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέτος και του χρόνου. Το Eurocore λοιπόν έχει αποδείξει ότι είναι απόλυτα δεσμευμένο για να συμμετέχει σε επιχειρήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το μόνο στρατηγείο που έχει τόσες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο φέρνοντας ε, πλήρως σε πέρας διάφορες επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Και τέλος περιμένουμε να παίξουμε το ρόλο του 2020 του Γενικού Στρατηγίου του NRF εφόσον βέβαια τα κράτη-μέλη μας θέλουν να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα ανα πάσα στιγμή μπορούμε να αναπτυχθούμε προς όφελος της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Όπως είπα και πριν, το Eurocore σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε ως στρατηγείο σώματος στρατού που μπορεί να κινητοποιήσει και να αναπτύξει έως και 65.000 στρατιώτες. Έχουμε το δικό μας στρατιωτικό δόγμα για να είμαστε χρήσιμοι στα πλαίσια της Ένωσης. Το Eurocore μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά κυρίως δίνοντας έμφαση όχι σε αποστολές ειδικά ε, μάχης, αλλά κατάρτισης για παράδειγμα για να εξοπλίσουμε και να καταρτήσουμε ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών αποστολές ε, βοήθεια στην άμυνα για να δώσουμε συμβουλές σε άλλες ένοπλες δυνάμεις, δημιουργίας στρατιωτικού δυναμικού, παρακολούθησης και ελέγχου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση της πληροφορίας και δομές ε, διοίκησης και ελέγχου στα πλαίσια αντιμετώπιση θεομηνιών ή κάθε είδους εκτάκτων καταστάσεων. Όλες αυτές οι αποστολές Βεβαίω ε, αποφασίζονται σε πολιτικό επίπεδο για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τις αξίες των εθνών και της Ευρώπης. Γι' αυτό θεωρώ ουσιαστικό να γνωρίζετε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει το Eurocore εάν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολή της Ένωσης. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις και οι δυνατότητές μας σε λειτουργικό επίπεδο είναι μια μοναδική ευκαιρία ούτω ώστε το Eurocore να έχει πιο στενές σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά τη γνώμη μου, ένα πιο υψηλό πολιτικό προφίλ του Eurocore στα πλαίσια της Ένωσης θα ήταν μεγάλο όφελος, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη του, αλλά γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε, ένα πρώτο βήμα έγινε 18 πρώτου, όταν υπέγραψα από πλευράς των πέντε κρατών μελών μία επιστολή προθέσεων με τον επικεφαλής του Γενικού Στρατηγίου Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε οι δύο οργανώσεις μας να συνεργαστούν. 18 Ιανουαρίου όπως είπα. Δηλαδή μόλις πριν λίγες εβδομάδες. Και το Eurocore επίσης είχε αναπτύξει το λεγόμενο κείμενο πλαίσιο, framework document, που δόθηκε στους αρμοδίους για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ε, Ένωσης. Τους εξηγούμε τι δυνατότητες έχουμε για να εκτελέσουμε τις αποστολές που προανέφερα πάντα προς όφελος της Ένωσης. Στις 2 προσεχούς Μαρτίου θα μιλήσω στην ε, Στρατιωτική Επιτροπή της Ένωσης για να τους εξηγήσω αυτό το κείμενο πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκα και νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Επιχειρούμε να το παρουσιάσουμε και σε άλλες πολιτικές ε, οργανώσεις και φορείς της Ένωσης της Βρυξέλλες. Αυτά βράχει πρόθεσμα. Μάκρο πρόθεσμα για να συμμετάσχει στους μηχανισμούς ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στο Eurocore πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική συμφωνία με τις ε, αρμόδιες αρχές της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη μας εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όπως είπα και πριν, στις 20 Απριλίου θα κάνουμε μία ε, διάσκεψη που λέγεται Post Allocation Conference όπου έχουν προσκληθεί όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης για να τους δώσουμε δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική πολυεθνική ευκαιρία ενός εμβρίου ευρωπαϊκής άμυνας. Όπως ε, καταλαβαίνετε το Eurocore έχει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Καταλήγοντας και πριν ε, σας μιλήσουμε ειδικά για την αποστολή μας στο Μαλί, τονίζω για να συνοψίσω ότι με δυνατότητες ε, διαταγών και ελέγχου το Eurocore μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου πολύ σύντομα. Χάρη στο ειδικό του καθεστώς και στον πλήρως, πλήρως και γνήσια πολυεθνικό του χαρακτήρα, το Eurocore έχει την αναγκαία νομιμοποίηση που είναι κλειδί της επιτυχίας του για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτή η πολυεθνικότητα. Βεβαίω ξέρετε, πολύ καλύτερα από μένα, η πολυεθνικότητα δεν σημαίνει πάντα απλές καταστάσεις. Μέσω εντόνων ε, ασκήσεων είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος ξεκινώντας με τη δημιουργία του σώματος μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ομάδας μάχης συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προσεχές εξάμεινο. Είμαστε δεθυμένοι για να αναπτυχθούμε σε οποιοδήποτε τύπου αποστολή ως ομάδα ακριβώς μάχης. Το Eurocore μπορεί να αξιοποιηθεί και μπορεί να είναι και το προτιμόμενο γενικό στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όποτε θέλετε, όπου θέλετε και ανεξάρτητα από την αποστολή που πρέπει να αναλυφθεί γιατί βελτιώνουμε τη συνεργασία μας. Την τέλειοποιούμε, όπως σας έλεγα, τη συνεργασία μας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στον ταξίαρχο κύριο Φρέγκλε ο οποίο ε, μόλις επέστρεψε από το Μαλί πριν από μερικέ εβδομάδε και θα σας μιλήσει συγκεκριμένα για την αποστολή μα στο Μαλί. Σα ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο ταξίαρχος Φρέγκλε. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους ήμουν ο επιτελάρχης της αποστολής EUTM ε στο Μαλί. Είναι αποστολή ε, που είναι διαδεδομένη με το ακρονίμιο EUTM. Βεβαίω υπάρχουν πολλέ αυτού του είδους στην κανονική μου ζωή, αν μπορώ να μιλήσω για αυτήν, είμαι του Eurocore, όπως το ανέφερε ο προλαλή σα. Όπως ξέρετε, η δική μας αποστολή στο Μαλί αποτελείται από δύο πυλώνες. Αφενός από τη συμβουλευτική ομάδα που βλέπετε κάτω αριστερά, Μιλάμε για περίπου 20 ιδιαίτερα πεπειραμένους αξιωματικούς στον Μπάμακο, αξιωματικοί οι οποίοι ε, παρέχουν συμβουλές ε, στο ε, Υπουργείο στο Μαλί. Είναι δηλαδή 20 άνθρωποι, λίγοι είναι, αλλά αυτοί όμως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και θα το εξηγήσω. Το δεύτερο που βλέπετε δεξιά είναι περίφημη Training Task Force. Πρόκειται δηλαδή για τους εκπαιδευτές των ε, δυνάμεων ενόπλων δυνάμεων του Μαλή που αυτοί είναι εγκατεστημένοι στο Κολικόρο περίπου 60 χιλιόμετρα από τον Πάμακο και κατά κανόνα ε, χρειάζονται δύο ώρες για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Της ε, αποστολής προείσταται ο επιτελάρχης στο Mission Headquarter Μπάμακο, 180 είναι εκεί οι στρατιώτες, η δύναμη αποτελείται από 180 άντρες. Αυτή λοιπόν η αποστολή είναι μια αμυγός ευρωπαϊκή αποστολή. Όταν ήμουνα στο Μαλί εκπροσωπούσα 23 κράτη και άλλα δύο τα 23 ήταν της Ευρώπης και τα άλλα δύο εκτός Ευρώπης γιατί είναι η μόνη αμυγός Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποστολή και πρέπει να σας πω ότι το Μαλί είναι ιδιαίτερα περήφανο που μπορεί να φιλοξενεί αυτή την αποστολή και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Η εντολή Παλκών 2 εφέτος ε, ισχύει η UTM κατά το τελευταίο εξάμεινο, εκτός από τις κανονικές εργασίες ε, της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης, έπρεπε επίσης να συμβάλλει ε, στην περίφημη στρατηγική αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Strategic Review. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο για την εντολή παριθμών 3 το αποτέλεσμα της εντολής 1 και 2 είναι πολύ θετικό. Μέχρι τώρα έχουμε εκπαιδεύσει 7 GTA Group Tactique ε, είναι μια στρατιωτική ε, δύναμη με 106 ε, άνδρες η οποία έχει τη δυνατότητα να ε, εκπαιδεύσει τις χερσαίες δυνάμεις. Και τα κατάφερε αυτή η GTAIA δύναμη γιατί κατόρθωσε να εκπαιδεύσει μάχημες δυνάμεις οι οποίες δίνονται και να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ε, κατάστασης. Τώρα, θα υπάρξει και άλλη μία όγδοη ομάδα μάχης η οποία από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να εκπαιδεύεται στο Κολικόρο. Έτσι λοιπόν στο τέλος της εντολής υπαριθμών 2 θα έχουν εκπαιδευτεί 8 ομάδες μάχης όπως ακριβώς προβλέπεται στην εντολή. Αυτές οι δυνάμεις κυρίε και κύριοι έχουν εκπαιδευτεί θαυμάσια με βάση αφρικανικά πρότυπα. Και κατ' ουσίαν αν θέλετε πρόκειται για την ελίτ, την αφρόκρεμα των δυνάμεων του Μαλή. Έχουμε λοιπόν 120 εκπαιδευτές οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί στο τέλος της εντολής και συνολικά ε, θα έχουν εκπαιδευτεί 7.500 άνδρες στο τέλος της εντολής. Παράλληλα με αυτό υπάρχουν και άλλες μικρές ομάδες στήριξης ε, που και με αυτές ε, ασχοληθήκαμε όσον αφορά την εκπαίδευσή, του, εκπαίδευσή τους. Τώρα, όσον αφορά την παροχή συμβουλών, η δύναμη EUTM συνέβαλε έτσι ώστε οι δυνάμεις ε, του Μαλή να έχουν ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη των δυνάμεων μέχρι το 1919. Αυτός ο νόμος ε, ε, έχει θεσπιστεί από το κράτος και η πρόκληση που υφίσταται είναι ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί με συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένη υποδομή. Και εδώ υπολείπονται πάρα πολλά. Αυτό που δεν πετύχαμε είναι το εξής. Με την εντολή υπαριθμών 2 να επιτύχουμε την δυνατότητα εκπαίδευσης ενόπλων δυνάμεων αποκλειστικά και μόνο από το Μαλί. Και αυτό οφείλεται στο ότι η εκπαίδευση των δυνάμεων του Μαλί, η εκπαίδευση αυτή έπρεπε καταρχήν να εστιαστεί σε συγκεκριμένες μονάδες για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση ή αν θέλετε για να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Στο μέλλον επιτρέψτε μου ε, να πω το εξή. Δεν θα είναι δυνατόν να διατηρήσουμε το συσταγωγικά εργοστάσιο μονάδων GTEA. Δεν θα γίνεται αυτό, δεν θα μπορεί να είναι δυνατόν. Θα πρέπει να αποσυρθούμε από αυτή την κατάσταση που είναι τώρα η ένοπλη σύνταξη σε μια μεταγενέστερη κατάσταση και εκεί να προκύψουν στρατιωτικά δόγματα και σχέδια έτσι ώστε οι ε, ένοπλες δυνάμεις του Μαλή να καταστούν αξιόμαχες. Στόχος λοιπόν είναι η σταθεροποίηση και με την εντολή υπαριθμών 3 αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα που πάλι σημαίνει ότι παράλληλα με την παροχή συμβουλών σε στρατηγικό επίπεδο πρέπει η παροχή συμβουλών να επεκταθεί και σε όλα τα άλλα επίπεδα και να περάσουμε από το στρατηγικό επίπεδο σε όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση του επιτελείου των αρχηγικών στελεχών εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, κατ' ουσίαν αυτό είναι το πρόβλημα των ενόπλων δυνάμεων του Μαλή. Δεν έχουν καλή καθοδήγηση. Και αυτό το αναγνωρίζει και ο Υπουργό και γενικότερα το επιτελείο, το στρατιωτικό επιτελείο στο Μαλή. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Η εκπαίδευση στα τάγματα θα πρέπει να βελτιωθεί γιατί δεν είναι αλήθεια ότι οι εκπαιδευμένοι μπορούν να έρθουν στο κολικόρ και να συνεχίσουν εκεί ε, την εκπαίδευση. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα από την εκπαίδευση με μεμονωμένων στρατιωτών αλλά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών έτσι ώστε οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλή να δίνανται, να αναλάβουν μόνες τους την εκπαίδευση. Μιλάμε λοιπόν για εκπαίδευση ταγμάτων τα στρατόπεδα. Μιλάμε λοιπόν για ε, επιχειρήσεις ε, προς ε, πολλών ε, οργανισμών ε, με στόχο την επίτευξη της ειρήνης. Για να τα επιτύχουμε όλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα συνεπές σύστημα, έναν κύκλο, έναν αποτελεσματικό κύκλο ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στο Μαλί στο πλαίσιο της ε, G5 Sahel να παίξει σημαντικότερο ρόλο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτή η νέα προσέγγιση που πραγματικά είναι αποκεντρωμένη αυτή θα συμβάλλει έτσι ώστε η δύναμη EUTM ε στο μέλλον να μην περιμένει τον πελάτη εισαγωγικά στο κολικόρο αλλά η ίδια να πάει στον πελάτη και η μονάδα αυτή να ξεφύγει από ad hoc προσωρινές στρατηγικές και μονάδες αλλά και μάλλον να προσαρμοστεί ε, στις ε, κανονικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Κατά την άποψή μου λοιπόν τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να πετύχουν καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων στο Μαλί και οφείλουμε να αναζητήσουμε καλύτερη συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις, με την αποστολή αυτή που εκπαιδεύεται και επιλαμβάνεται των αστυνομικών δυνάμεων. Μινούσκα και Μπακάμε θα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο και ε, νομίζω ότι ε, μπορούμε να παίξουμε ε, συμπληρωματικό ρόλο επιτόπου. Εν κατακλείδη κυρίες και κύριοι, η εντολή 3 και η εφαρμογή της από του χρόνου ε, από το Μάιο του επόμενου χρόνου ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλει έτσι ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας καλύτερα την εκπαίδευση αρχηγικών στελεχών. Και η παροχή συμβουλών θα επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε αποκεντρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Βήμα προς βήμα δεν είναι βέβαια δυνατόν να τα επιτύχουμε όλα το Μάιο, θα προχωρήσουμε σταδιακά γιατί η αποκέντρωση έτσι κι μπορεί να επιτευχθεί μόνο σταδιακά. Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξω είναι ότι θέλουμε ε, να βοηθήσουμε το Μαλί να βελτιώσει, όπως σας είπα, τους εκπαιδευτές σε αρχηγικό επίπεδο και την αποτελεσματικότητά τους. Αλλά πάντα έχοντας κατά νου τα στάνταρτ της Αφρικής. Δηλαδή δεν θα επιδιώξουμε το ανώτατο δυνατό επίπεδο. Ε, δεν θα ε, μπορέσουμε να επιτύχουμε όλα αυτά που ισχύουν για τις ε, ισπανικές και γερμανικές ε, στρατιωτικές δυνάμεις. Πάμε τώρα στο εξής. Ποια είναι τα πλονεκτήματα που έχουν προκύψει. Αφενός το ότι υπάρχει καθημερινή συνεργασία σε διεθνές πλαίσιο. Δηλαδή ισχύει το εξής. Ένας αξιωματικός από μια ευρωπαϊκή χώρα που δούλεψε στο επιτελείο, ο <clears throat> αξιωματικός αυτός δεν είχε εργαστεί ποτέ σε πολυεθνική ε, υποδομή και μου είπε, ξέρετε εμείς σκεφτήκαμε ότι α, έρχεται το Eurocore και ε, κανένα πρόβλημα, αυτό και μόνο φτάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ε, ήρθε το Eurocore, αλλά συνεχίστηκε η καθημερινότητα σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό το να ενταχθούν δηλαδή οι γηγενείς σε αυτό το πλαίσιο και αυτό ε, θεωρώ ήταν πολύ σημαντικό. Εμείς λοιπόν όπως σας είπα προσφέραμε το επιτελικό προσωπικό το να μπορεί λοιπόν κανείς σε αυτή τη φάση να συμβάλλει στην αποστολή και να καταθέσει προτάσεις για το μέλλον αυτό ήταν σημαντικό και ήταν σημαντικό επίσης να υπάρχει προσωπικό του Eurocore επιτόπου. Γιατί το προσωπικό αυτό έχει συνηθίσει να σκέπτεται όχι μόνο στο κατώτατο αλλά και στο ανώτατο επίπεδο. Και πρέπει να ξέρετε ότι ανάμεσα στον επιτελάρχη του ΕΟΤΕΜ και του ΠΕΣΚΑ δεν υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνο ο πρόεδρος ε, της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο διοικητής ε, πρέπει να καλύπτει όλα τα επίπεδα και χρειάζεται το απαραίτητο επιτελείο να τον στηρίζει. Τι πέτυχε το Eurocore. Πρέπει να σας πω ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Συγκεντρώσαμε εμπειρία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ενδεχομένως και άλλες ένοπλες δυνάμεις. Συγκεντρώσαμε εμπειρία και από την Αφρική και μας ε, ενδιαφέρει επίσης και η άμεση συνεργασία με διάφορους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί <clears throat> και η διαδικασία Αθήνα-Αθήνα. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Σε γενικές γραμμές λοιπόν κυρίες και κύριοι Κατά την άποψή μου ε, αυτή η αποστολή ήταν μια θαυμάσια προετοιμασία για το Eurocore, για να μπορεί το Eurocore να αναλάβει και άλλες επιχειρήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνάδελφός μου ήδη αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές ομάδες μάχης, τα battle groups. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Okay, I'm going to open. Uh, can we ask uh, Dan John. Excuse my pronunciation. Ο, ο κύριος John. Ζητώ συγγνώμη για την ε, προφορά μου. Καλημέρα σας ε, και καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε για τις εξαιρετικά πλήρεις εισηγήσεις σας. Αρκετοί εξημών ήδη γνωρίζουμε το Eurocore και θα πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που χαιρετίζω σήμερα μια ιστορική σημασία πρόοδο του Eurocore, δηλαδή την ολοκλήρωση μιας αποστολής προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ε, ο τίτλος Ευρωπαϊκό Σώμα, Eurocore, πολλές φορές έχει οδηγήσει σε λάθος αντίληψη, ε, καθώς πολλοί πίστευαν ότι πρόκειται για, εξ αρχής για μια δομή που ήταν συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ, όπω είπατε, στρατηγέ, ποτέ δεν είχατε εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε λοιπόν τη χαρά μα που αυτή τη φορά το Eurocore ε, επιτέλεσε μια αναποστολή προ όφελο τη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ε, και ε, ε, επίσης με χαροποιεί το γεγονός ότι είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό ε, μέσω των Battle Group, των ομάδων μάχης 150 όπως είναι γνωστές αλλά και με τους υπόλοιπους τρόπους που μας αναλύσατε και που μπορείτε να παρέμβετε. Μιλήσατε για πολλά ζητήματα που έμεναν σε κρεμότητα οπότε δεν έχω πραγματικά ερωτήσεις αλλά ήθελα απλά να υπογραμμίσω ότι ανάμεσα στα ισχυρά σημεία επί των οποίων επιμείνατε φυσικά ο πολυεθνικός χαρακτήρας ε, του, της δομής η διτή αυτή η προσωπικότητα ο ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αλήθεια πως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί δυστυχώς να υπάρχει μια καχυποψία ε, από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, από στρατητική άποψη. Εξακολουθούν κάποιες χώρε να είναι φοβισμένες και να λένε καλύτερα να πάμε με, από το ΝΑΤΟ, με το ΝΑΤΟ. Εγώ πιστεύω πως αυτό είμαστε συμβατοί. Ε, θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το γεγονός ότι το EuroCorp μπορεί να κάνει ένα σωρό αποστολές ε, μαζί με την ε, δύναμη γρήγορης αντίδρασης του ΝΑΤΟ, έχοντας τον ευρωπαϊκό αυτό χαρακτήρα, μπορεί αυτό να καθησυχάσει όλο τον κόσμο. Οπότε δίνει ένα χαρακτήρα ε, ενταξιακό θα έλεγα για όλους, ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να εισχωρήσουν και άλλες χώρες. Και τρίτο πλεονέκτημα της Eurocore ήταν ότι απέδειξε και αυτή η αποστολή η UTM Μαλή το απέδειξε αυτό. Η εκπαιδευτική αποστολή της Ένωσης στο Μαλή απέδειξε και έχετε πολύ αφοσιωθεί σε αυτή την αποστολή και μάλιστα ε, ήρθατε και μας ενημερώσατε κάθε φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποδείξατε τις δυνατότητες του Eurocore που θεωρούσε, θεωρήθηκε αρχικά όταν πολύ μεγάλο και πολύ εξελιγμένο για να ασχοληθεί με μικρές ευρωπαϊκές αποστολές. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι σε θέση να το κάνει μέσω αυτής της αποστολής στο Μαλί. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες αποστολές στο μέλλον, ε, αποστολές ε, πολλές και διάφορες, ε, εκπαίδευση, συμβουλή, πλαισίωση, ακόμα και ε, αποστολή μάχης, πάντως το Eurocore μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις αποστολές και στα όλα τα ίδια αποστολών. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή. Ε, θα συνεχιστούν οι ανταλλαγές απόψε. Θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε και μεμονωμένα τα μέλη αυτής της υποεπιτροπής για να μπορέσετε να τους πείσετε για τη χρησιμότητα της δομής ε, του Eurocore και για την ευελιξία που προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής άμυνας της για το μέλλον της Ευρώπης είναι αυτή η ευελιξία. Μιλήσαμε για έννοιες, για πιο δογματικές δομές. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα μέσω της ευελιξίας και το EuroCorp προσφέρει αυτή την ευελιξία σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καρποφόρες ανταλλαγές απόψεων στο θέμα. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. Ο κύριος Φροντζουλίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο στρατηγούς για τις εισηγήσεις τους. Κυρίε και κύριοι, θυμάμαι πριν από πολύ καιρό όταν ε, Δημιουργήθηκε το Eurocore το 1992. Εργαζόμουν στις εξωτερικές υποθέσεις Ρουμανίας και ήμουν υπεύθυνο για το ΝΑΤΟ και τη Δυτική ε, Ευρώπη. Και αυτή η ιδέα που προέκυψε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να δημιουργήσουν το Eurocar κατά κάποιο τρόπο συνδέθηκε με τις δυτικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και τώρα θεωρείται έτσι. Και έτσι λοιπόν θεσπίστηκε αυτό το ανεξάρτητο σώμα και πραγματικά ήλπιζα ότι αυτό το Eurocore τελικά θα μπορούσε να αποτελέσει το αρχικό την αρχική βάση για μια πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη άμυνας και ασφάλειας. Ε, δεν θέλω να επικρίνω τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πραγματικά ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει το Eurocore ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δομών της. Δυστυχώς παρέμεινε πάντοτε μια μικρή στρατιωτική δυνατότητα ένα μικρό θεσμικό σώμα που παρέχει υπηρεσίες στις χώρες που συμβάλλουν στην συντήρησή του. Ταυτόχρονα, στη διάρκεια αυτών των 23 ετών, το Eurocore ε, είχε μόνο τέσσερις σημαντικές αποστολές. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να δούμε με τις ευρωπαϊκές χώρες κατά πόσο το Eurocore θα μπορούσε να ενισχυθεί γιατί με αυτές τις δυνάμεις δεν μπορεί να ασκήσει πραγματικά ειρηνευτικές αποστολές αλλά μόνο να ανταποκριθεί σε αποστολές χαμηλής έντασης. Να δούμε λοιπόν με τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά πόσο μπορούμε να χτίσουμε πάνω στο Eurocore μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατιωτική δομή. Διότι δυστυχώς κυρίες και κύριοι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα σωρό απειλές για τη σταθερότητά της και την ασφάλειά της που έτσι όπως έχει τώρα που είναι μια ήπια δύναμη δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Ίσως θα πρέπει να ε, ε, οικοδομήσουμε λοιπόν πάνω στη Eurocore μια πιο ε, μεγάλη δύναμη, πιο ισχυρή δύναμη για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις απειλές. Μάλλον, κατά τη γνώμη μου, και αυτό θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η δική σας γνώμη, κατά πόσο, δηλαδή, αν οι ευρωπαϊκές χώρες αποφασίσουν να ενσωματώσουν το Eurocore στις ευρωπαϊκές δομές αμήνης, αν θα μπορούσατε, όπως προτείνατε κάποτε, να γίνεται ε, μια δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη αντίδρασης. Όλοι φοβούνται βέβαια να μην τυχόν γίνει επικάλυψη με τον ΝΑΤΟ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βασίζουν την ασφαλειά τους και την άμυνά τους στο ΝΑΤΟ για την ώρα και όχι σε ευρωπαϊκές δομές. Το Eurocore βέβαια ακόμα και τώρα βασικά αντιπροσωπεύεται από την γαλλογερμανική ταξιαρχία. Εξαιρετικό παράδειγμα. Αλλά σε 23 χρόνια θα έπρεπε πάνω σε αυτό να έχουν χτιστεί κι άλλα. Ωστόσο η Eurocore εξακολουθεί να είναι μια πολύ μικρή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, Mr. Uh, ευχαριστώ κύριο Γιούρακ. Ευχαριστώ πολύ. και να ευχαριστήσω και τους δύο αξιωματικούς για τις σημαντικές τους παρουσιάσεις. Ιδιαίτερα για τη δραστηριότητα του Eurocore. Ένας προηγούμενος ε, σας ρώτησε για τις προοπτικές του Eurocore. Ξέρω ότι από την αρχή ε, στόχος του Eurocore ήταν ακριβώς να αναπτυχθεί να εξελιχθεί. Να εξελιχθούν οι δομές του και να συνδεθεί με τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεργασία, να συνεργαστεί και με τα όργανα της Ένωσης και με το ΝΑΤΟ, γιατί χρειαζόμαστε μια αμυντική πολιτική και ο καλύτερος τρόπος ε, να την αποκτήσουμε είναι να επιδείξουμε αλληλεγγύη στα πλαίσια της Ένωσης και να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ. Διερωτώ λοιπόν, θα είναι δυνατόν το Eurocore να είναι το όργανο άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνατότητες κοινών ασκήσεων. Ασκήσεων στρατιωτικού αμυντικού χαρακτήρα, όχι απλώς ε, κατάρτιση, όχι απλώς εκπαίδευση. Θα ήταν δυνατόν το Eurocore να κάνει τέτοιες ασκήσεις στις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξωτερικής απειλής για να ενισχύσουμε την αμυντική ικανότητα κάποιων κρατών μελών. Αναφέρομαι κυρίως ε, στα ανατολικά της Ένωσης φυσικά. Θεωρείτε ότι τέτοιες δραστηριότητες ε, έχουν έννοια. Θα ήταν χρήσιμες γιατί ξέρω ότι έχετε ήδη πείρα από τέτοιες ασκήσεις. Θα ήταν δυνατόν λοιπόν να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες. κυρία Βότμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, γνωρίζω το Eurocore Ε, Επισκέφθηκα για δύο μέρες κατά μία ολομέλεια πέρυσι το Eurocore και θυμάμαι τις ε, εξηγήσει που μου δόθηκαν και τις προφορίες και εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ που οργάνωσα άλλη μία ε, επίσκεψη που θα γίνει στις 10 Μαρτίου με συναδέλφους από την ομάδα μου, τη φιλελεύθερη ομάδα ALDE. Μας εντυπωσιάζει πολύ η δραστηριότητά σας και πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο το Eurocore. Διότι έχουμε πολλά γεγονότα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ένταξη της Πολωνίας και αυτήν την ε, δήλωση προθέσεων στις 18 Ιανουαρίου μεταξύ του ε, Γενικού Επιτελείου της Ένωσης και του Eurocore που προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών και μια σειρά από όλες τις δραστηριότητε. Και μετά μιλήσατε και για την αποστολή στο Μαλί. Και όσον αφορά αυτή την δήλωση προθέσεων, χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η προσέγγιση μεταξύ του EuroCorp και του στρατιωτικού επιτελείου της ε, Ένωσης ε, ως μέλος φυσικά της Επιτροπής ΕΝΤΕ. Και όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, εξετάζουμε ένα κείμενο για την συνεργασία μεταξύ της ασφάλειας και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί σε αυτές τις ε, περιόδους κρίσης δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πρέπει να συνεργάζονται οι δημόσιες αρχές με ιδιωτικούς φορείς και αυτό μπορεί να γίνει και στον τομέα της ε, άμυνας και της ασφάλειας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό. Ξέρω ότι το στρατηγείο σας, για παράδειγμα, ε, απασχολεί μια ιδιωτική υπηρεσία για την ασφάλειά του. Άρα τι μπορείτε να μας πείτε περισσότερο για αυτό τώρα, για το Μαλί. Κάνατε πολλά για την κατάρτιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αυτής. Ξέρω ότι η αποστολή αυτή πήγε καλά αλλά ποια είναι τα διδάγματα που έχετε εξαγάγει από αυτή σας την αποστολή και πώς θα αξιοποιήσετε αυτά τα διδάγματα στα πλαίσια των μελλοντικών σας ε, αποστολών εκπαίδευσης ενόπλων δυνάμεων γιατί πρέπει να συμμεριστούμε αυτή σας την πείρα και κάτι για πώς βλέπετε τις προπτικές σας που πιστεύω ενδιαφέρει και πολλούς άλλους συναδέλφους. Πολλοί εξακολουθούν να λένε το Eurocore είναι ο στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι νομίζουν πολλοί έτσι, όταν ε, συζητούμε μαζί τους. Ο πρόεδρος Σούλτς πριν από μερικά χρόνια είχε μιλήσει για ευρωπαϊκές ενόπλες δυνάμεις. Ποια είναι η δική σας θεώρηση. Θεωρείτε το Eurocore θα μπορούσε να γίνει αυτό ο στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι ορισμένοι προσδοκούν μια τέτοια εξέλιξη. Θα θέλατε να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς το ρόλο σας σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους ε, της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ένωσης. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, κυρίως μας απασχολεί η κρίση ασύλου και μετανάστευσης. Είναι η σημαντικότερη πρόκληση στην παρούσα συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι πολίτες μας γνωρίζουν ότι για να επιληθεί αυτή η κρίση πρέπει να βρούμε λύσεις που να μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε τον έλεγχο των συνόρων μας. Το συζητήσαμε και χθε. Και μας εξέπληξαν κάποιες ε, απαντήσεις που λάβαμε. Θέλω να μας πείτε τι ρόλο θα μπορούσατε να παίξετε σε αυτό. Θεωρείτε ότι μπορείτε να έχετε κάποιο ρόλο, μπορείτε να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη στον καλύτερο έλεγχο των συνόρων της Ένωσης. Το έχετε σκεφτεί αυτό καθόλου. Εάν θέλουμε να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους μας και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα τις απόψεις σας. Η κυρία Βαλρό. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω σου ειδικά τη στιγμή που μου προσφέρετε σήμερα αυτή η δυνατότητα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το 2008 ε, πήγα στο Μαλί πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και τότε το Μαλί ήταν ε, ήδη μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου όπου γινόταν αισθητή η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή υπήρχαν πολλά προβλήματα για τους ανθρώπους επιτόπου. Ε, θα έπρεπε τότε ήδη να αλλάζουν τις μεθόδους καλλιέργειας. Εγώ λοιπόν πήγα στο Μαλί για να δω μόνη μου πώς λειτουργεί η αναπτυξιακή πολιτική της ε, Σουηδίας. Το Μαλί λοιπόν είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν να εγκαθιδρυθούν δημοκρατικά συστήματα στη Δυτική Αφρική. Σε άλλες ε, χώρες ε, πολλοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να μιμηθούν το παράδειγμα του Μαλή. Βεβαίως και υπάρχουν στη χώρα διάφορες πολιτικές ομάδες ε, και αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις που σιγοβράζουν. Σε μια δημοκρατία όμως ε, είναι γεγονός ότι ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος των συγκρούσεων. Είναι μια χώρα η οποία όπως σας είπα γίνεται όλο και πιο φτωχή και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανοίγει διάπλατα την πόρτα για το ενδεχόμενο των συγκρούσεων. Το ίδιο βιώσαμε και στη Λιβύη. Εσείς λοιπόν είσαστε επιτόπου εκεί και άλλοι πηγαίνουν επί τόπου στο Μαλί. Μας ε, είπατε ότι συνεργαζόσαστε με την αστυνομία για να είναι η αστυνομία μάχημη σε ε, περιπολίες. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες που βρίσκονται στο Μαλί έτσι ώστε η χώρα να μετατραπεί σε ειρηνική μια χώρα όπου να μπορεί κανείς να εργαστεί όπως εργάζονται όλοι, να είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις ε, της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά που σας λέω τρέχουν παράλληλα. Και θέλω να ρωτήσω, υπάρχει άραγε κάποια μορφή συνεργασίας με άλλες ε, ομάδες της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών ή με τις πρεσβείες που εκπροσωπούνται, που βρίσκονται επί τόπου, συνεργάζεστε με αυτούς. Γιατί μερικές φορές ισχύει το εξής, οι στρατιωτικοί δεν συνεργάζονται απαραίτητα με τους πολιτικούς εθελεντές. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός, όμως η κατεύθυνση πρέπει να είναι κοινή. Κύριε Σεφχάουζερ. Σας ευχαριστώ πολύ για τι παρεμβάσει. Θέλω να κάνω τρει παρατηρήσει. Η πρώτη αφορά την ιδιαιτερότητα του Eurocore. Είστε ένα όργανο που συστήθηκε από δύο κράτη, τη Γαλλία και τη Γερμανία στην αρχή. Μετά επεκτάθηκε χάρη στη βούληση της Γαλλίας και της Γερμανίας με στόχο την ενισχυμένη συνεργασία και την ανεξαρτησία. το όραμα του κυρίου των κυρίων Μητεράν και Κολ ήταν να συστήσουν μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή δύναμη άμυνας. Γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος ύπαρξής σας. Υπάρχει το ΝΑΤΟ. Γιατί να γίνει το Eurocore αν δεν υπήρχε αυτή η ανεξαρτησία. Και ακριβώς αυτό με κάνει τη δεύτερη μου παρατήρηση. Εάν χάσετε την ανεξαρτησία σας, εάν κανείς σας συγχαίει με το ΝΑΤΟ, δεν έχετε πλέον λόγο ύπαρξης. Άρα λοιπόν, πρέπει να διατηρήσετε αυτή την, αυτό το όραμα ανεξαρτησία. Και μάλιστα μετά την πτώση του τείχους και την πρώτη συνεδρίαση του Βίζεγκραντ ήμουν στην ε, ε, πηγή. Μιλήσαμε για αυτήν την εξαρτησία. Η Ευρώπη ήταν έτοιμη. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης ήταν έτοιμες για την ανεξαρτησία στην, στην αμυνά τους. Αλλά δυστυχώς, και θα πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, δεν είχαμε τα μέσα για να στηρίξουμε την ανεξαρτησία μας. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως ο προπολογισμό θα αυξανόταν και θα είχαμε δηλαδή τα κοινά μέσα, βεβαίως, τα οποία δεν έχουμε όμως. Και πιστεύω πως θα πρέπει λοιπόν να διδρύσετε αυτή τη σας και δεύτερον την ανεξαρτησία σας και κατά τρίτο λόγο να μείνετε σε αυτό το προφίλ, σε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση, σε μια καμπή πολύ ουσιαστική της Ευρώπης. Η Ευρώπη όπως την είχαμε ε, αντιληφθεί ε, και συλλάβει εξ αρχής την Ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν λειτουργεί πλέον. Τι λειτουργεί η Ευρώπη των Εθνών, της συνεργασία, η Ευρώπη που ενδεχομένως να έχει διάθεσή τις διάφορες πολλαπλές δομές όπου θα υπάρχει προσθέμενη αξία και σε αυτό το όραμα μπορείτε να το διατηρήσετε με την προϋπόθεση ε, βεβαίω να διατηρήσετε και επαναλαμβάνομαι ίσως, συγγνώμη, να διατηρήσετε αυτή την εξαρτησία που ήταν η ιδιωτική πράξη μιας ανεξάρτητης Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστείτε με το ΝΑΤΟ. Η Γαλλία, η χώρα μου, ανέκαθεν όταν χρειαζόταν ήταν με την πλευρά του ΝΑΤΟ. Αλλά καταρχάς ήταν ανεξάρτητη. Και ξαλώ το λέω συχνά και στους Πολωνούς φίλους μου, δεν πρέπει να τρέφουν αυταπάτες. Εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για την άμυνά μας, δεν θα μας υπερασπιστεί κανείς. Και τέλος, τελευταία παρατήρηση για ένα στοιχείο που μου είχε διαφύγει, η Τουρκία. Δεν γνώριζα ότι ήταν δεμένο μέλος η Τουρκία. Ειλικρινά, αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Πρέπει να είμαι ε, ειλικρινής απέναντί σας. Σήμερα το μέγα πρόβλημα των μεταναστών και των όσων γνωρίζουμε δεν είναι το πρόβλημα των μεταναστών που καταφτάνουν. Μπορώ να το καταλάβω. Και ότι θέλουν να δεθούν το καταλαβαίνω. Για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα ή για να ε, επιβιώσουν. Το οργανωμένο έγκλημα που διαχειρίζεται τις ροές των μεταναστών ε, με ποσά που φτάνουν τα 9 με 10 δις ε, αυτό αποφέρει η διαχείριση των μεταναστών στα οργανωμένα αυτά κυκλώματα. Το πρόβλημα ότι η Τουρκία ε, στην Τουρκία λειτουργεί το αλβανικό οργανωμένο έγκλημα και εφόσον έχετε ένα σύστημα πληροφοριών θα γνωρίζετε περί τίνος πράγματος μιλάω. Πώς θέλετε λοιπόν να συνεργαστείτε και να διαχειριστείτε μια ανεξάρτητη Ευρώπη απέναντι στο μεγαλύτερο, αυτή, στη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει με την Τουρκία που παίζει ένα τελείως αντιευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να το ξεκαθαρίστε αυτό για το μέλλον σας, γιατί διαφορετικά δεν θα έχετε μέλλον. Και πιστέψτε με, εμένα που πιστεύει σε αυτή την Ευρώπη των κρατών, την Ευρώπη των εθνών, την Ευρώπη της συνεργασίας, εάν εσείς αποτύχετε στο στόχο τους, δεν θα έχει μέλλον ούτε η Ευρώπη, γιατί η Ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν λειτουργεί. Εάν δεν λειτουργεί ούτε η Ευρώπη των εθνών, ε, τότε ειλικρινά δεν ξέρω. Χάνω τον μπούσουλα. General ε, Με κάθε σεβασμό, ε, στρατηγέ μου, Φρέγκλε, διαφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε ότι έχουμε μονάδες απόλυτα εκπαιδευμένες που τις αποκαλείται ε, μονάδες ειδικών δυνάμεων. Προφανώς πρέπει να εφαρμόσουμε αφρικανικά πρότυπα και στάνταρ. Αλλά έχω πείρα και ξέρω ότι τα αφρικανικά πρότυπα σε ορισμένα μέρη όταν εφαρμόζεται μια φράση του ισπανικού ύμνου του πεζικού όταν ξέρεις να πεθάνεις, ξέρεις και να νικήσεις που δεν είναι ρητορική, είναι πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οι, γαλλικές, ε, η γαλλική λεγεώνα των ξένων καταστράφηκε από αντάρτες και αντιμετώπισαν όλοι αυτοί κανόνες στο Φάντα, κανόνια συγγνώμη, στην Φάντα και το Γουαντιντούμ και καταστράφηκαν ακόμη και μονάδες που υπεράσπιζαν τη βάση του Ματαντσάρα του Συμφώνου της Βασοβίας. Το θεμελιώδες και το ξέρετε εσείς που είστε στρατιωτικοί πρέπει να είναι στρατιωτικές μονάδες που να είναι διατεθειμένες να πεθάνουν. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο Μαλί. Στο Μαλί η σταθερότητα εγκαταστάθηκε, επανήλθε χάρη στην ε, ε, ε, επιχείρηση Μπαρχάν. Χάρη στις δυνάμεις ασφαλείας και τις δυνάμεις πληροφοριών και τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που εκμεταλλεύτηκαν τις αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων εθνών και φυλών. Ορισμένες από αυτές τις φυλές ε, εξοπλίζονται από τη Γαλλία. Τι γίνεται επί τόπου. Κάποια στιγμή οι μονάδες που ήταν διτεθειμένε να σκοτώσουν και να πεθάνουν, που ήταν ε, οι απόλυτα αποτελεσματικές δυνάμεις ενός απόλυτου ε, ενός απόλυτα εκπαιδευμένου στρατού, του στρατού του Τσάντ, αυτές νίκησαν. Εγώ ήμουν στο Μαλί. Κατά τη θητεία του στρατηγού Γκαρθία Βακέρο. Και γύρισα τρομοκρατημένος και τρομοκρατημένος το λέω ήπια. Γιατί η εντολή που έχετε είναι μια εντολή ευνουχισμένη. Και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Φταίμε εμείς, οι πολιτικοί. Εσείς ξέρετε αυτό που σας λέμε κάνετε, αυτό που σας λέμε να κάνετε. Αλλά οι μονάδες του EUTM λένε ότι δεν είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουμε επιθετικά, αλλά μόνο αμυντικά τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαν να είμαστε στο μεσαίωνα όταν είχαμε φρούρια και καθόμασταν πάνω στα τείχη και τα υπερασπιζόμεθα. Το ξέρετε πολύ καλά. Σε κάθε πόλεμο τώρα και ιδίω σε πόλεμο ερήμου, για να μπορέσει κανεί να αμυθεί σε βάθο, σε ανοιχτέ περιοχέ, δηλαδή 350-400 χιλιόμετρα ελέγχου, και όταν υπάρχουν ε, στο, όπως στο Τεσσαλίτο και στο Κιδάλ ορεινές περιοχές που τις γνωρίζω, όταν πρέπει να αμυνθούμε εκεί, πρέπει να καταστρέψει οποιαδήποτε μπει σε αυτό το, στην περίμετρο ασφάλειας. Αλλά βεβαίω αν κάνεις ε, επιθετικές επιχειρήσεις τότε πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ε, πεθάνουν ή να υποχωρήσουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια στρατιωτική επιθετική ε, επιχείρηση ο λόγος απολειών είναι τρία προς ένα και ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιστράφηκε αυτός ο, αυτός ο λόγος στις επιθέσεις που κάναμε εκεί. Γιατί όλα αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία. Πρώτον, η εκπαίδευση είναι απόλυτα μη αποτελεσματική. Μετά από τρία χρόνια εκπαιδεύσεως δεν έχουμε ειδικέ δυνάμεις, δεν έχουμε λειτουργικές δυνάμεις και μονάδες καμία δυνατότητα ε, να επιχειρήσουν. Γιατί δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα, δηλαδή δυνατότητα να επιχειρήσουν. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε επιτόπου για να αποτιμήσουμε τι δυνάμει έχουμε. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, εξαρτώμεθα από αυτά που θα μας ε, διηγηθούν. Δεν μπορούμε εμεί να αποτιμήσουμε τι δυνάμει έχουμε και τι δυνατότητες έχουν να επιχειρήσουν. Δεύτερον, ο οπλισμός του, Επειδή είμαστε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφυσική και φιλοσοφική, ο οπλισμός πρέπει να είναι του στρατού του Μάλι. Δεν του δίνουμε λοιπόν επιθετικό υλικό. Γιατί ξέρουμε ότι είναι κακή ανατροφή να σκοτώνει τον εχθρό σου. Του εκπαιδεύουμε, ελπίζοντα ο στρατό του Μαλή θα του δώσει την επιθετικότητα που χρειάζεται. Το μόνο που είχε η e UTM ήταν δύο όλμοι ε, των 60 χιλιοστών. Και ούτε LPR-7 δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γιατί δεν υπήρχε ε, το κατάλληλο υλικό. Δεν είχαμε όπλα 14,5, δεν είχαμε το PU-23. Αυτά είναι βασικά όπλα δεν είχαμε DBM21, δηλαδή τα ε, όργανα του Στάλιν, που έχουμε αυτές τις στοιχείες πυράβλων. Μα τι ενέχουν αυτά όταν ε, ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε δυνάμεις ιδιαίτερης κινητικότητας. Ενώ αυτά τα όπλα είναι όπλα για κορεσμό πυροβολικού σε περιορισμένη περιοχή. Σας το λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει εκπαίδευση. Γιατί δεν γίνεται επιθετική εκπαίδευση, δεν υπάρχει αποτίμηση εκπαίδευση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η σχέση μεταξύ ε, στρατιωτών και αξιωματικών είναι η χειρότερη. Είναι τόσο κακή κατάσταση, και ξέρω γιατί λέω, είναι τόσο κακή κατάσταση που οι αξιωματικοί ε, δίνουν εντολέ και διαταγέ από τα μετόπισθεν. Οπότε και οι στρατιώτε ε, δεν πολεμούν, διότι αν δεν έχουν μαζί του αξιωματικούς φυσικά την κουπανάνε. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Και τρίτον, ξέρετε ότι η κατάσταση των φυλών σε όλες τις αφρικανικές χώρες οι, οι κάτοικοι του Νότου, οι Μπαμπαρά, οι του Κολέρ δεν ενδιαφέρονται καθόλου να πάνε να πεθάνουν στο Βορρά που είναι τύπος εδάφους που δεν γνωρίζουν παρά το ότι μεταφυσικά είναι στην ίδια χώρα. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οι νητές του Άρες, Μόρα, Σόγκα και Πεούλ. Επίσης η Γάτιας, βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες ε, μονάδες από αυτές τις φυλές. Δημιουργούμε λοιπόν πολλοί βραδικίνητες μονάδες που δεν μπορούν να πολεμήσουν σε αυτό τον πόλεμο κίνησης. Κοιτάξτε, όταν για παράδειγμα ο βασικός τρόπος μετακίνησης είναι ορισμένα φορτηγά ή κέντρα ανεφοδιασμού, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάποια, κάθε μονάδα ξέρει ότι για να υπάρχει ε, κινητικότητα χρειάζεται τα κατάλληλα οχήματα. Ο στρατός του Τσάντ έχει το Ιώτα. Κάθε το Ιώτα έχει και ε, νερό, έχει και φαΐ και έχει και ξύλα για να ανάβει φωτιά. Όλοι οι στρατιώτες ε, τρώνε μαζί, δεν εξαρτώνται από κάποιον να τους φέρει τρόφιμα. Δεν εξαρτώνται από ένα όχημα το οποίο μπορεί να έχει καταστραφεί το μεταξύ ή να έχει χαλάσει και δεν φτάνει. Πώς είναι δυνατόν τόσο βαριές μονάδες στην έρημο χωρίς να έχουν τε, ε, σκηνές. Αυτό είναι σαν να σκεφτόμαστε... Α, συγγνώμη, δεν χρειάζονται σκηνές. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να τις στήσει και μετά πρέπει να την ξεστήσει. Και αν έχει αέρα θα πέσει. Γιατί γίνει το χειρότερο εχθρό σου. Γιατί θα πεθάνεις εκεί πέρα μέσα όταν πέσει πάνω σου. Και ένας πέθανε. Γιατί του έπεσε πάνω η σκηνή ή ε, τα παλούκια της σκηνή και το σκότωσαν. Αυτά τα ξέρουν όλοι όσοι πολεμούν στην έρημο τι δημιουργούμε. Μονάδες οι οποίες δεν παίζουν κανένα ρόλο. Και ο οπλισμός τους είναι οπλισμό οπλισμός ελαφρύς. Δεν είναι κατάλληλο, δεν είναι προσαρμοσμένο. Και κάθε φορά που πολεμήσαμε τους Χέτια, την κοπάνησαν τρέχοντας. Δεν λειτουργήσαν. Δύο χρόνια εκπαίδευση θα έπρεπε να αρκέσουν για να ε, δημιουργήσετε μονάδε. Οι μονάδε οι οποίε εκπαιδεύτηκαν από το γαλλικό στρατό στο Σαλάλ εκπαιδεύτηκαν σε 40 μέρες αλλά είχαν επιθυμία να αγωνιστούν, είχαν επιθυμία να πεθάνουν γιατί αγωνίζονταν για τα εδάφη τους. Ο στρατηγός Γκαρθία Μακέρο μου είπε κάτι που με εξέπληξε και με έκανε να γελάσω. Μου είπαν ότι θα εκπαίδευαν μονάδες και ελπίζω να μην έγινε αυτό για να εκπαιδευτούν κοντά στα ποτάμια και για να μπορούν να διασχίσουν ποτάμια. Αλλά κοιτάξτε, στην περιοχή που θα πολεμήσουν δεν έχει ποτάμια. Πάνω από τον ποταμό Νιζέρ. Είναι πολύ περίπλοκο να περάσει κανείς ποτάμι. Είναι ενδιαφέρον. Αλλά αυτά είναι σαν να τους λέτε στην Γρυλανδία πώς θα πρέπει να πολεμήσουν στην έρημο. Γιατί? Για τις ε, επιχειρήσεις ειρήνης μου είπαν. Αλλά αφού όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα γίνουν στο βορρά. Δηλαδή εκπαιδεύουμε μονάδες που είναι απόλυτα άχρηστες. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Και ο Μαμπαντού ρε, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, μου είπε, κοιτάξτε, χρειαζόμαστε μονάδες από το Τσάντ. Και εσείς μας εκπαιδεύετε με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στα ισπανικά λέμε ότι η κίνηση αποδεικνύεται όταν κινείται κανείς. Και εδώ και τρία χρόνια είμαστε σταματημένοι. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι Πρέπει να απαντήσετε, πρέπει όμως να τελειώσουμε στις 10.30. Θα αφήσω να αποφασίσετε μεταξύ σας ποιος θα απαντήσει σε ποια ερώτηση. So, ε, bueno, ε, ε, Να σχολιάσω, τις δια... είχε, υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και αυτό πολύ με ευχαριστεί γιατί σημαίνει ότι σας τραβήξαμε την προσοχή, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα πρώτο στόχο που επετεύχθη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ή, εν πάση περιπτώσει, να σας εκφράσω τη σκέψη μου για τις πολλές ερωτήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν ε, ερωτήσεις αλλά σχόλια ή συμπεράσματα. Και θα προσπαθήσω στα πέντε λεπτά να απαντήσω. Όντως, η Eurocore, έτσι όπως έχει φτιαχτεί, και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το Eurocore είναι ε, ένα ανεξάρτητο σώμα και είναι αυτό που επιθυμούν τα κράτη-μέλη του να είναι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό, αυτή η διτή σχέση με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνθημα του Eurocore είναι Eurocore μια δύναμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΝΑΤΟ. Και για τον ΝΑΤΟ λέει από την αρχή. Ε, συστήθηκε το Eurocore για διάφορους ε, και πολλούς λόγους. Από το 1998 πάντοτε κάναμε αποστολές για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2015 ήταν η πρώτη φορά που ήταν καθαρά αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια αλλαγή, αυτό βλέπω και εγώ, και πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή και να μετατρέψουμε σε πραγματικότητα αυτό το σύνθημα, αυτό το τη ρίση που χαρακτηρίζει το Eurocorp για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ. Τώρα, είπατε, αποτελεσματικότητα και ευελεξία. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Πρόκειται για μια στρατιωτική δύναμη που αποτελείται από 55.000 ανθρώπους. Ναι, Σκέφτεται κανείς ότι είναι μεγάλα τα άγματα αυτά, αλλά δεν ισχύει αυτό πλέον. Δεν ισχύει ότι είναι μεγάλη η δύναμη αυτή. Εμείς κινούμαστε όντως στο χώρο της ε, ευελιξίας. Και είναι αλήθεια ότι όταν ο Κόλ και ο Μιτεράν ε, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Eurocore, σκέφτονταν την Ευρωπαϊκή Άμυνα, δεν σκέφτονταν τον ΝΑΤΟ. Αυτό που είναι πάντως βέβαιο είναι ότι το Eurocore μετετράπει στο πρώτο ε, στο πρώτο βάση, στην πρώτη βάση, στο πρώτο τούβλο το οποίο, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ναι, Στρασβούργο, Ευρωπαϊκή Δύναμη, θα πρέπει πάντα να εξηγούμε ότι είμαστε στο Στρασβούργο, ναι, αλλά το Eurocore δεν είναι η Ευρωπαϊκή Πολεμική Δύναμη, ε, ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Είμαστε λίγο παραπάνω, αντιπροσωπεύουμε λίγο παραπάνω από τις μισές χώρες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πάντως, η οι κύριοι αυτής της στρατιωτικής δύναμης είναι αυτές οι 5-6 χώρες. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Eurocore εργάζεται για τα έθνη, για τα έθνη framework, όχι. Εκείνοι είναι λοιπόν οι κύριοι, ε, τα αφεντικά. Αλλά εργαζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ. Δεν εργαζόμαστε στι εσωτερικέ αποστολέ τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ισπανία, του Βελγίου κτλ. Είπαμε ότι είναι διπλό ο χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ. Για το μέλλον τώρα του Eurocor Και κατά πόσο πρέπει να υπάρχει κάποιο είδο συμμαχία με το ΝΑΤΟ. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια ε, έχει υποθεί. Και θα πρέπει ειλικρινά να σας το πω. Δεν υπήρχε κανένα χαρτί, κανένα έγγραφο όπου να υπάρχει ρητά ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στο Eurocore και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα απολύτως, μηδέν, πουθενά δεν αναφερόταν αυτό. Ξεκίνησε αυτή η σχέση με την υπογραφή του επιστολής συνεννόησης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το EuroCore. Eurocorp τώρα. Και αυτό όντως ε, προετοιμάζει το μέλλον. Είναι ένα βήμα για το μέλλον. Ένα άλλο θέμα, το θέμα των προσφύγων και τι μπορεί να κάνει το Eurocorp. Τι να σας πω σήμερα, ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, τα θέματα Ασφάλεια και αμυνα πανε πάνε χέρι-χέρι. Παλαιότερα υπήρχε μια σαφή διάκριση. Λέγαμε αυτό είναι θέμα άμυνα, το άλλο είναι θέμα ασφάλεια. Τώρα είναι αλληλένδετα. Σχεδόν δεν υπάρχει πλέον διαφορά. Έχουμε βέβαια τις γαλλικές ενόπλες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή έχουν την επιχείρηση Sentinel φρουρός που προσπαθεί να αυξήσει την ασφάλεια με ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ενόπλων δυνάμεων στις δρόμους των πόλων, το ίδιο και στο Βέλγιο. Τώρα, τι ρόλο μπορούμε εμείς να παίξουμε για το θέμα των προσφύγων σήμερα. Εγώ, ως επικεφαλής του Eurocorp δεν έχω καμία απολύτως εντολή, καμία σχέση με το θέμα των προσφύγων. μέσα σε αυτό το, εντάσσεται μάλλον περισσότερο στο θέμα της ασφάλειας και όχι της άμυνας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορεί αύριο να αλλάξουν πάντως, τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχω καμία σχετική εντολή. Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Eurocorp. Είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία. Πέντε κράτη. Και ε, εντός ολίγου και η Πολωνία. Είναι λοιπόν τα πέντε κράτη, συν, ε, συντόμως έξι, τα κράτη-μέλη της ε, Europol. Έχουμε συνδεδεμένα μέλη, συνδεδεμένα κράτη, που έχουν δηλαδή χτυπήσει την πόρτα της EuroCorp και, να, και έχουν πει μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με αυτό το EuroCorp». Αλλά δεν ε, συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις είπαμε ε, ε, δεν είναι, δεν είναι αξιωματική, δεν μπορεί να συμμετέχουν σε κάποιες φάσεις σε ασκήσεις. Αυτό είναι όλο. Η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση σε απόρριτες πληροφορίες που αφορούν μόνο τα ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε συμμετέχει στο Battle Group. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσω εντό πέντε λεπτών, υπήρχαν και πολλά ερωτήματα για το μαλλί. Και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να απαντήσω. Ίσως το, πάντως το μόνο σαφές μήνυμα που θα ήθελα να σας διαβιβάσω είναι το εξής. Αυτή η διάσκεψη για την καταχώρηση των θέσεων είμαι πεπισμένος ότι το Eurocore είναι ένα σώμα που έχει μέλλον είναι κατά κάποιο τρόπο το έμβριο ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού στρατού Η Ευρώπη χρειάζεται ευρωπαϊκό στρατό. Ήδη εμεί αντιπροσωπεύουμε πάνω από το ίμιση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πάντω, έτσι όπω έχουν τώρα τα πράγματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να, αυξηθεί, να αυξηθούν οι δυνάμει του Eurocorp. Πάντω, η νομιμότητα ε, έχει σχέση με την, τον πολυεθνικό χαρακτήρα. Πέντε συν μία χώρες. Προσεχώς θα είμαστε έξι γιατί αυτός ο πολυεθνικός χαρακτήρας σημαίνει ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε στον Ευρωπαϊκό Στρατό. Στις 20 Απριλίου θα γίνει εδώ θα γίνει εδώ μια διάσκεψη καταχώρησης ε, θέσεων και θα θέλαμε να ανοίξουμε σε περισσότερες χώρες ε, συνδεδεμένα κράτη, οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα δεν είναι μέρο και θέλει να συνδεθεί είναι ευπρόσδεκτο εννοείται και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ομιμότητα και τον πολυεθνικό χαρακτήρα του Eurocore. Αυτά, τίποτα άλλο, ε, έρχεται έχετε το λόγο. Meine Damen und Herren, es wird mit Sicherheit nicht... Κυρίες και κύριοι, δεν θα σας εκπλήξει βέβαια το ότι θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Νατ. Κύριε Βουλευτά, θα μου άρεσε πάρα πολύ να είχα τη δυνατότητα να πιούμε μαζί ένα βράδυ εδώ στο Στρασβούργο ένα καλό ε, ποτήρι ισπανικό κρασί και να τα πούμε. Ε, σας κερνάω κιόλας και νομίζω ότι θα βρούμε αυτή τη δυνατότητα να τα πούμε και φαντάζομαι εκεί ε, πραγματικά θα έρθουμε σε ουσιαστική αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, απευθύνομαι στον άλλο κύριο, εγώ δεν είπα ότι στο Μαλί είναι όλα καλά, ε, που δεν είδε ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Επίσης, για μένα δεν τίθεται το θέμα κατά πόσο μπορούμε να προετοιμάσουμε τις ε, ένοπλες δυνάμεις του Μαλί για επιθετικές ε, ή για μηντικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι τους εκπαιδεύσαμε για κάτι που μπορούν να κάνουν, κυρίως για θέματα ασφάλειας και σταθεροποίησης. Επίσης, ε, ίσως ε, δεν ξέρω μπορεί να σας άρεσε όρος που χρησιμοποίησα ή αφρόκρεμα αλλά ξέρετε η λέξη αυτή ισχύει για τα τοπικά πρότυπα γιατί αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί από εμάς είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ε, απειλές στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων. Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της χώρας. Θα το πω έτσι λίγο άγαρμα, ε, το να δει κανεί αν κάποιος είναι μαχητής ή όχι, πολεμιστής ή όχι. Είναι κάτι σημαντικό αυτό. Μετά, ε, συνοδεία και στήριξη. Αυτό επίση είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίμαχο όπως γνωρίζετε. Νομίζω όμως ότι τώρα πια με τον αναπροσανατολισμό των επεμβάσεων ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση των στελεχών. Και πράγματι η ε, ικανότητες των αξιωματικών και των υπαξιωματικών αν δεν βελτιωθούν οι αρχικές τους ικανότητες νομίζω ότι θα αποτύχουμε. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω και κάτι χαρακτηριστικό από την εκπαίδευση. Ήμουνα στο Κολικόρο στην εκπαίδευση και εκεί είχε γίνει το εξής, ε, ε κάποιοι ε, άντρες έπεσαν σε ενέδρα και μετά το συζητήσαμε αυτό. Ένας λοιπόν πολύ καλός αξιωματικός ήταν στο πρώτο αμάξι, στο πρώτο όχημα του κονβόι, μετά ακολουθούσαν άλλα και μετά όταν το συζητήσαμε εκ των υστέρων είπα ε, στον αξιωματικό που ήταν επικεφαλής ε, Πού ήσουν εσύ, εγώ ήμουν στο τελευταίο όχημα και του λέω μα πώς είναι δυνατόν ένας αξιωματικός στο τελευταίο όχημα και του λέω Κοίταξε να δει. το γεγονό ότι ο αναπληρωτή σου ήταν στο πρώτο όχημα, αυτό ήταν καλό, αλλά εσύ έπρεπε να είσαι το πολύ στο δεύτερο. Γιατί ο αξιωματικό είναι εκείνο που καθοδηγεί, δεν είναι εκείνο που απλά πλαισιώνει και στηρίζει. Και επίση να σα πω ότι ε, το είπα αυτό και στον αρχηγό του κράτους και στου άλλου αξιωματικού. Δηλαδή πρέπει να θέσουμε βάσεις στι φρουρές. Αν δεν δημιουργήσουμε τα θεμέλια δεν μπορούμε να τις αναβαθμίσουμε αυτές τις φρουρές και να τις καταστήσουμε battle groups. Αυτό που παίζει ρόλο είναι αυτή η προσπάθεια. Και το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί και η αξιοπιστία ε, των ενόπλων δυνάμεων στα μάτια των ίδιων των κατοίκων της χώρας, αυτό νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Ελπίζω ε, να ήταν κατοπιστικά αυτά που είπαμε. Όπως σας είπα, σας καλώ να τα πούμε ένα βράδυ και ευχαρίστω να συζητήσουμε σε βάθος. Επιτρέψτε μου να φέρω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Ε, ο Ρουμάνος συνάδελφός σας έθιξε το θέμα της συνεργασίας. Κατά την άποψή μου το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο έχει συνηθίσει να ηγείται διαφόρων εθνικών ομάδων. Γιατί ε, ποτέ δεν θα είναι σαφές ευθύς εξ αρχής ε, ποια ομάδα θα συμμετέχει σε ποια αποστολή. Και μιλάμε για ένα επιτελείο το οποίο επίση έχει συνηθίσει να συνεργάζεται με του θεσμού Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι ενωσιακέ διαδικασίε. Αυτό δεν μπορεί κανεί να το μάθει μέσα μία μέρα. Αυτό στο Μαλί εγώ το έμαθα ε, έξι μήνε κάθε μέρα και αυτή είναι μία ανεκτήμητη εμπειρία που πρέπει να τη μεταφέρουμε και στους υπολείπους. Τώρα όσον αφορά την ε, εκπαίδευση Πράγματι εμείς ε, εξασκούμεθα για το FHQ Battle Group και προβαίνουμε στην εκπαίδευση των ανδρών. Μετά όμως θα ε, ασχοληθούμε και με την εκπαίδευση ε, που θα αφορά την NATO Response Force. Το ερώτημα σχετικά με τη μετανάστευση. Είναι σαφές ε, ότι ο διοικητή που προηγήθηκε τα είπε όλα πολύ σωστά. Μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι του Μαλή αγαπούν τη χώρα τους. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μείνουν εκεί, στη χώρα τους. Κατόπιν τούτου οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Αλλά ξέρετε κυρία Βαλέρο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μια κατάσταση ασφάλειας, αν είναι ικανοποιητική η ασφάλεια, ε, επιλύονται κατά κάποιον τρόπο κατά κάποιον τρόπο τα άλλα προβλήματα. Όμως να το πω αλλιώς ότι αν δεν υπάρχει ασφάλεια οξύνονται τα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Άρα δηλαδή ε, αυτά τα δύο θέματα όπως σας είπα, αυτά που έδειξα και αυτό που λέω τώρα συμβαδίζουν. Η, ο συντονισμός γίνεται κάθε εβδομάδα ακόμα και στο πλαίσιο της ε, αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μάλι και θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός ο συντονισμός όταν θα μεταβούμε επιτόπου στις διάφορες περιφέρειες και θα προβούμε στην αποκέντρηση. Εκεί επιτόπου κατάλαβα ότι η συνεργασία ανάμεσα στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τι πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στρατιώτες είναι τόσο καλή που ποτέ δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και τους δύο στην Επιτροπή μας που μας ενημερώσατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας, μας βοηθήσατε πάρα πολύ και θέλω να σημειώσω ότι σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για μας και επίσης σας ενημερώνω ότι οι επόμενες δύο συνεδριάσεις μας είναι στις Βρυξέλλες 17 και 18 Φεβρουάριο. Πέρα συνεδρίες. Ευχαριστώ πολύ.